Dear colleagues. συνάδελφοι. Είναι μεγάλη χαρά να συναντάτε ανθρώπους από ξένες επιτροπές. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ λίγο. Σήμερα θα κάνω μια ανταλλαγή απόψεων με την, τον Παγκοσμίο Οργανισμό Τροφίμων για την κατάσταση των τροφίμων στον κόσμο. Έχουμε πάρει μία αίτηση για να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και τα, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων Χαίρομαι που έχουμε τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΔΕΒΕ και την Επιτροπή Άγκρη που ήρθαν και αυτοί για την συζήτηση κοινή και πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως δίνον τον λόγο για σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις στους συναδέλφους μας πρώτη η κυρία Μακέβαν Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Είχαμε ε, μια συνέντευξη της Επιτροπής μας και ξεπεράσαμε το χρόνο μας όπως κάνουμε πάντα. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την κοινή συζήτηση εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων την Παρασκευή. Είναι μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Έχουμε μια σημαντική έκθεση η οποία θα μας παρουσιαστεί. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να είναι κανείς από την πείνα και είναι ένα τμήμα των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας. Ο στόχος ήταν να μειώσουμε στο μισό τον αριθμό των ατόμων που πλήττονται από την πείνα στο 2015. Έχει επιτευχθεί αυτό, αλλά είναι ακόμα 795 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο που πεινάνε. και το μισό των ε, θανάτων των παιδιών κάτω από 5, πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο, οφείλεται στην, ε, στον υποσυτισμό. Στο παρελθόν το έχουμε παραγνωρίσει το θέμα αυτό στα προγράμματα μας του 80 και του 90. Δεν δώσαμε αρκετή έμφαση στην, σε επενδύσεις στη γεωργία και την τροφιμική ασφάλεια. Αυτό ξεκίνησε να αλλάζει στο τέλος της τελευταίας δεκαετίας, αλλά θα πρέπει να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο οι στόχοι ανάπτυξης της χιλιετίας εκπνέουν την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και θα διατυπωθεί τότε το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης για τα επόμενα 15 χρόνια. Δύο εβδομάδες ε, πριν στη Νέα Υόρκη συναντήθηκαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών του κόσμου και όλοι έχουν δεσμευτεί για νέους παγκόσμιους στόχους. Ένα από αυτού είναι ο στόχος ανβιώσιμη ανάπτυξης 2, είναι να επιτύχουμε το τέλος της πείνα, να αυξήσουμε την ασφάλεια τροφίμων και να προωθήσουμε τη βιώσιμη γεωργία. Ως πρόεδρο τη ε, επιτροπή ε, <clears throat> Ανάπτυξης και εσείς και οι άλλες επιτροπές, όλοι μα είμαστε δεσμευμένοι να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να συνεργαστούμε την Κομισιόν και να ελέγξουμε τα κράτη-μέλη μας για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Τέλος. Δεν μπορεί κανείς να έχει τρόφιμα χωρίς γη. Η πρόσβαση στη γη είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που η Επιτροπή Αναπτυξή μας θα πάει στο Μιλάνο στο τέλος της εβδομάδας, στην Expo 2015 για να συζητήσει για τα θέματα της τροφιμικής ασφάλειας και την Πέμπτη το βράδυ, το απόγευμα, θα έχουμε μια ειδική συνάντηση, ένα εργαστήριο της Επιτροπής Ανάπτυξης για το θέμα της πρόσβασης στη γη, ανθρώπινα δικαιώματα και ασφάλεια τροφίμων στο Μιλάνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που με καλέσατε εδώ και προσβλέπω στην συνέχεια αυτό που θα πείτε για την έκθεση. Τώρα ο Πρόεδρος Ετζέσκη, Πρόεδρος Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας είναι μια μεγάλη διεθνής πρόκληση και έχει πολλές σημαντικές πτυχές. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές πτυχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Διεθνής Οργανισμός ε, Τροφίμων ζητά να μπορέσουν τα κράτη του κόσμου να βρουν συστημικές λύσεις για να ξεπεράσουν τα προβλήματα της ένδυας, της πείνας και του αποκλεισμού κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε πολύ καλές εμπειρίες με όλα αυτά τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια αγροτική πολιτική που έχει εξασφαλίσει και έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα, τις τελευταίες δεκαετίες και νομίζω ότι αυτές οι εμπειρίες θα μας βοηθήσουν να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά τα θετικά παραδείγματα και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε μια κοινή πορεία σε ό,τι αφορά την ε, ανάπτυξη και το εμπόριο με τις χώρες του τρίτου κόσμου μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπόριου οι πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβουμε θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα εξαλειφθεί η, η πείνα. Πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη αλλαγή στις χώρες αυτές του τρίτου κόσμου ώστε να πάψει να υπάρχει η πείνα. Δεν θέλουμε να κάνουμε μοναχα καλοπιστικές αλλαγές με τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνουμε έχουν να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω και την κρίση των προσφύγων. Είμαστε επομένως υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι αντί να ζητούμε και βρίσκουμε παγκόσμιες λύσεις και λαμβάνουμε υπόψη και τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν για περισσότερη έρευνα η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και φυσικά η έρευνα αυτή θα βρει συγκεκριμένη εφαρμογή στις χώρες όπου οι άνθρωποι πεινούν ακόμα και εν κατακλείδη θα ήθελα να αναφερθώ στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον αγροτικό τομέα και με το περιβάλλον. Είναι αποφασιστικό σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και το, τα λοιπά, να τα κάνουμε και στον τομέα της γεωργίας και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή τροφίμων. Κάτι ακόμα που θέλω να τονίσω όταν μιλάμε για διατροφή, αυτό είναι αποφασιστικό, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της, ε, των υδατίνων πόρων. Για να έχουμε μια υγιή διατροφή είναι απαραίτητη η σωστή υδατινή πόρη και αυτό είναι μια μεγάλη αξία για όλους μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον πρόσωπο του ΦΑΟ, τον κ. Μουσταφά Μνασέρ, ο οποίος είναι διευθυντής στο ΦΑΟ, liaison officer με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυρία Κριστίνα Πετνάσκα που είναι ε, διευθύντρια του προγράμματος για το είδο εδώ στις Βρυξέλλες. Θα δώσω το λόγο για 10 λεπτά στον καθένα και μετά θα αρχίσει η συζήτηση μεταξύ μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης και σας που οργανώσατε αυτή τη συζήτηση για να μιλήσουμε για το διατροφικό ζήτημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η εβδομάδα που γιορτάζουμε την ε, Παγκόσμια ημέρα για τη διατροφή. 16 Οκτωβρίου. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία για να προβληματιστούμε όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια ανά τον κόσμο. Να σκεφτούμε τα θέματα λοιμού, τα θέματα ένδυας στην Ήπεθρο και να δούμε τι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως είπε και η κυρία Μακάβεν. Να δούμε τι γίνεται με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ο στόχος 2 ε, αναφέρεται στην ε, απάλληψη της φτώχειας. Συνεπώς, η προσπάθεια είναι μια κοινή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους παράγοντες για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Στο ΦΑΟ θεωρούμε ότι η απάλληψη της φτώχειας το 2030 είναι ένας ε, στόχος εφικτός, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, αρκεί να θέσουμε στη διάθεσή μας ε, τα μέσα που έχουμε. Στην έκθεση του Μιλάνου πράγματι θα γίνουν εκδηλώσεις με εκπροσώπηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι ευκαιρία για να συνεχίσουμε την συζήτηση για αυτό το καυτό ζήτημα. Εποφέλουμε από την ευκαιρία εδώ για να σας πω επίσης ότι σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του ΦΑΟ ξεκίνησε με την έκθεση ΣΟΦΑ που είναι ουσιαστικά για την κατάσταση όσον αφορά για την διατροφή και τη γεωργία σε ολόκληρο τον κόσμο. Την έκθεση αυτή από το 1947 κάθε χρόνο την εκπονεί ο ΦΑΟ. Και είναι κάτι που βοηθάει βέβαια τι πολιτικέ αποφάσει, του πολιτικού δηλαδή για να πάρουν πολιτικέ αποφάσει. Η έκθεση αυτή λοιπόν φέτο για την κατάσταση τη γεωργία και των τροφίμων ανά τον κόσμο επικεντρώθηκε κυρίω στο ρόλο τη κοινωνική προστασία στα πλαίσια της καταπολέμησης της ένδυας και της πείνας ε, μέσω της προώθησης της ανάπτυξης της υπαίθρου και της γεωργίας. Δέκα λεφτά μας δώσατε, οπότε θα, αναφερθώ, θα αναφέρω μόνο κάποια κέρια μηνύματα. Σήμερα ξεκίνησε και το site για αυτά τα ζητήματα. Τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας οδηγούν στη μείωση της ένδυας και του υποσυτισμού εποφελούνται όλοι. Βέβαια οι βοήθειες πρέπει να προσαρμόζονται και είναι βασικό στοιχείο αυτό για την επιτυχία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα θέματα αυτά έχουν ε, περισσότερες επιπτώσεις πάνω στις ε, γυναίκες που υποφέρουν περισσότερο. Τα θέματα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε και να υποστηρίξουμε περισσότερο τους πιο δύναμους. Να δούμε και τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά την ε, παραγωγή τροφίμων. Ε, να δούμε την παιδεία που μαζί με την ένδια και τον υποστητισμό επηρεάζουν το μέλλον των ανθρώπων. Η κοινωνική προστασία όμως από μόνη της δεν φτάνει για να απαλληφθεί η πτώχεια. Τα πιο φτωχά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ένα σώρο περιορισμούς και κινδύνους. Γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε σε κοινά προγράμματα, συντονισμένα, ώστε να συνδέσουμε την κοινωνική προστασία με τη γεωργία. Και όλα αυτά βασισμένοι σε πολιτικές και στρατηγικές που υιοθετούν οι διάφορες χώρες. Οι δράσεις μας μαζί με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής, είναι να στηρίξουμε τέτοιες χώρες. Και θέλω να αναφέρω εδώ ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με τη βοήθεια της ΔΕΦΚΟ, για να βοηθήσουμε ακριβώς τις χώρες να εθετήσουν πολιτικές και στρατηγικές για την καταπολέμηση του υποσυτισμού. Τέλος, η κοινωνική προστασία έχει θετικές επιπτώσεις σε κοινότητες και οικονομίε σε τοπικό επίπεδο. Ε, τα δημόσια έργα μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές και πόρους συλλογικούς, άρα να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία. Τέτοια βοήθεια στηρίζει και τα νοικοκυριά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τέτοια έργα. Σήμερα πολύ χαίρομαι που έχω μαζί μου εδώ έναν συνάδελφο που ασχολείται με τη διατροφική ασφάλεια, αλλά και τη συνάδελφο του ΠΑΜ, όπως είπατε και εσείς. Γιατί το ΠΑΜ, το ΦΙΝΤΑ και ο ΦΑΟ, και οι τρεις στη Ρώμη, συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους της επιστημιστικής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, εσείς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, με μεγάλη χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την έκθεσή μας για την επισητιστική ασφάλεια στον κόσμο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η έκθεση αυτή από το 1999 κάθε χρόνο υποβάλλεται και είναι μια κοινή έκθεση που ετοιμάζει ο ΦΑΟ με το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας είναι δηλαδή κοινό πρόγραμμα των τριών υπηρεσιών της Ρώμης που ασχολούνται με την επιστηστική ασφάλεια στον κόσμο. Η φετινή έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία. Το 2015 είναι σημαντική χρονιά για όλους μας, γιατί μας φέρνει στο τέλος ενός κύκλου. Τι σημαίνει αυτό? Από το 1996 ξεκινήσαμε με τους ε, επικεφαλείς κατά κυβερνήσεων που συναντήθηκαν στην Ρώμη το 2019 και φέτος με την δήλωση της χιλιετίας και με τον πρώτο στόχο είπαμε ότι όσον αφορά τον υποσυτισμό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ότι πρέπει να μειώσουμε κατά το ίμιση τον υποστισμό από το 1990 μέχρι το 2015. Είμαστε κοντά στην επίτευξη των ε, στόχων της χιλιετίας. Το στόχο δηλαδή όσον αφορά τον ε, υποσυτισμό, την πείνα. Είναι το ποσοστό που μας είπε να ελέγξουμε η διεθνή κοινότητα. Βλέπουμε λοιπόν στις αναπτυγμένες περιοχές ο δείκτης αυτός από το 23% πήγε στο 29%. Αυτό σημαίνει ότι στατιστικά είμαστε κοντά στην επίτευξη του στόχου. Οι 73 από τις 129 αναπτυσσόμενες χώρες που ελέγχονται για αυτή την περίοδο έχουν πετύχει το στόχο. Όμως, εδώ πρόκειται για ένα ποσοστό των πεινασμένων μέσα στο συνολικό πληθυσμό. Υπήρχε όμως και ένας άλλος στόχος που ήταν η μείωση του αριθμού των ατόμων που υποφέρουν από υποσυτισμό. Είναι ο στόχος της διάσκεψης για τη διατροφή και δεν είμαστε πολύ μακριά από την επίτευξη του στόχου. Θα έπρεπε να είχαμε μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των επισητιζόμενων. Όμως δεν είναι υπερβολικά αρνητικό αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά την περίοδο ελέγχου αυξήθηκε κατά 2 στα 2 δισεκατομμύρια ο πληθυσμός στον κόσμο. Άρα πολύ δύσκολο να επιτεθεί ο στόχος. Πάντως 29 χώρες επιτεύθηκε από τις 129 δηλαδή που ελέγξαμε. Άρα υπάρχουν κάποιες επιτυχίες. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι υποσυτισμένοι. Φυσικά στην έκθεση υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά εδώ έχετε μια συνολική εικόνα, όπου βλέπετε ότι στην Νότια Ασία έχουμε τον ε, μεγαλύτερο αριθμό υποσυτιζόμενων και το μεγαλύτερο ποσοστό και ακολουθεί η υπό Αφρική. Είναι η περιοχή επίσης όπου το φαινόμενο είναι περισσότερο παρόν. Οι ποσιτιζόμενοι είναι δεύτερη στη σειρά, αλλά σαν αριθμό είναι περισσότεροι και στην Νότια Ασία. Ποιοι είναι τώρα οι παράγοντες εκείνοι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και που οδηγούν σε επιτυχία. Ξέρουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη σίγουρα αποτελεί κινητήριο δύναμη για να μειωθεί ο υποσυτισμό. Αλλά πρέπει να συμμετέχουν όλοι στην οικονομική ανάπτυξη και να έχουν όλοι ευκαιρίες. Επίση, αύξηση της παραγωγικότητας, κυρίως των μικροπαραγωγών. Η κοινωνική προστασία είναι ένα τρίτο στοιχείο, πολύ βασικό, βάσει του οποίου πέτυχαν πολλές χώρες. Είναι όμως σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τη λειτουργία των αγροτικών ε, αγορών. Ποιο είναι το σύστημα διεθνούς εμπορίου, τι ωφέλη προσφέρει και να προσέξουμε και τις χώρες όπου υπάρχει κάποια κρίση και να προλαμβαίνουμε τις κρίσεις. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο αργά, λέει ο πρόεδρος. Ε, προσπαθούσα να πετύχω το χρόνο μου γι' αυτό. Κοινωνική προστασία, λοιπόν, την είπαμε για να προλαμβάνουμε κρίσεις. Πράγματι, σε τέτοιες ε, χώρες όπου υπάρχει κρίση, ο υποσυτισμός είναι πιο έντονος. Τέλος, ποιες είναι οι προοπτικές μετά το 2015. Είμαστε στο, είμαστε στο τέλος ενός κύκλου παρατήρησης και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε μπροστά μας μία ατζέντα για βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνουν διάφορους στόχους μέχρι το 2030. Η διεθνής κοινότητα ήδη δουλεύει σκληρά προκειμένου να πετύχει στόχους και δείκτες. Σημαντικό είναι εδώ να υπογραμμίσουμε ότι ο ποσιτισμός θα έχει εξέχουσα θέση. Είναι ο δεύτερος στόχος, αλλά θα υπάρχουν και άλλοι που θα πρέπει να παρατηρήσουμε και πολύ περισσότερα στοιχεία πάνω στα οποία να δουλέψουμε από πλευρά δικτών. Πρέπει να γίνει επίση πολλή δουλειά για να βελτιώσουμε και την τεχνολογία που διαθέτουμε για να ελέγξουμε τους δείχτε αυτούς σε διάφορε χώρε. Εδώ θέλω να αναγνωρίσουμε ότι η DEFCO μας έδωσε μεγάλη στήριξη τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο αυτό. Έχουμε προγράμματα για την παρατήρηση της πείνας στον κόσμο με νέους δείκτες για, την, ε, για τον επόμενο κύκλο παρατήρησης. Είναι τεράστια προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Yeah. Ναι, ε, okay. κύριε Πρόεδρε, ε, των, κύριε Πρόεδρε των Επιτροπών, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ε, δυνατότητα που έχω να λάβω το λόγο ενώπιόν σας. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να λάβω το λόγο ενώπιόν σας. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για να σκεφτούμε καλύτερα την πρόοδο, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά και τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας οι συνάδελφοι του ΦΑΟ σας έχουν παρουσιάσει την ε, έκθεσή τους με συγκεκριμένες προτάσεις για τους μηχανισμούς οι οποίοι θα πρέπει να υλοποιηθούν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με πιο γοργούς ρυθμούς τους, ε, την πρόοδο που πρέπει να απαιτείται. Τα στοιχεία, τα αριθμητικά είναι αστρονομικά, 800 εκατομμύρια ανθρώπων υπό το φάσμα της πείνας. Αλλά πίσω από όλα αυτά τα στοιχεία, τα αριθμητικά, υπάρχουν ανθρώπινα δράματα, παιδιά, τα οποία χάνουν τη ζωή τους. Εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε για όλους αυτούς. Έχουμε κάνει πολλές επισκέψεις στην Ιορδανία, όπου είδαμε οικογένειες προσφύγων, που πλήττονται και αυτοί από το φάσμα της πείνας. και μας έδωσαν να καταλάβουμε πόσο αδύναμοι νιώθουν που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα πια με τα παιδιά τους. <clears throat> δεν έχουν τη δυνατότητα να θρέψουν πια τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να παίξουν πια το ρόλο των γονέων και να δώσουν στα παιδιά τους τα στοιχειώδη πράγματα που απαιτούνται. Και είναι πολύ σπάνια ο πατέρας μας με την οικογένειά του γιατί πρέπει όλη τη μέρα να ψάχνει να βρει κάτι για να φάνε τα παιδιά του. ...650 ε, δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι τα χρήματα τα οποία δαπανώνται και σπαταλώνται... ...ενώ πολλά παραπάνω, πολλά από αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν την ε, πείνα. Έχουμε ένα τεράστιο πολιτικό και οικονομικό αλλά και ηθικό πρόβλημα. 40% των ε, αναγκών των ε, προσφύγων της Συριακής κρίσης, μόνο 40% μπορούν να καλυφθούν από το ΦΑΟ. <clears throat> Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε οδυνηρές επιλογές, να μειώσουμε στο ίμιση τις μερίδες τη διατροφής για τους πρόσφυγες και Επίσης γνωρίζουμε και αυτή η προβληματική έχει συζητηθεί πολλές φορές στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ο κόσμος έχει αντιμετωπίσει εφέτος ένα τεράστιο αριθμό εκτάκτων ανθρωπιστικών δράσεων σε παγκοσμίο επίπεδο που απίτησε πρόσθετους ε, πόρους όπως η κρίση του, της έμπολα, κρίση στο Ιράκ, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τον ΕΠΑΡ κτλ. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει υποστηρίξει όλες αυτές τις ενέργειες η πρόσφατη <coughs> επίσκεψη του, της κυρίας Μακάβαν, του κυρίου Ζέλερ και άλλων, έχουν, είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν το έργο, το έργο μας σε ένα καταβλισμό ε, προσφύγων. Εμείς ε, βοηθούμε 40.000 ε, πρόσφυγες της, της Συρίας εκεί. Συνεργαζόμαστε επίσης και με τους συναδέλφους της ΔΕΦΚΟ, του ΦΑΟ και άλλες κυβερνήσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τα προβλήματα αυτά, τα διαφορετικά της πείνας και, ε, και του υποσυντισμού. Μας ενώνει ο στόχος να εκπηδενήσουμε την πείνα στον κόσμο σε, στα επόμενα δέκα χρόνια. Θέλουμε λοιπόν να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πολλές φορές δυστυχώς οι έκτακτες κρίσεις ξεσπάνε εκεί όπου η κατάσταση τροφιμικής ασφάλειας ήταν ήδη επισφαλής, κάτι που εκθέτει τον, πολ, τον πληθυσμό σε ένδια, πείνα αλλά και ευαλωτότητα όπως γίνεται στο, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο Μαλί και σε άλλες χώρες που πλήττονται από την Εμπόλα οι αρχέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει σημαντικές προσπάθειες να δώσουν μια έκτακτη οικονομική βοήθεια στις χώρες αυτές και να εξασφαλίσουν και μια ανθρωπιστική βοήθεια προς τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για το γεγονός ότι οι αρχέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναφέρει τι προσπάθειε μα ω κύριε συνιστώσεις της επίλυσης της Συριακής κρίσης. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι το ΠΑΜ και η συνεργάτες μας συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις κοινέ προκλήσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε ευρώ το οποίο έχει δοθεί από τους Ευρωπαίους πολίτες με το πιο διάφανο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρουντόλφε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ αξιότιμη προεδρεύοντες, Πρόεδρε των επιτροπών, εξότιμοι ευρωβουλευτές. Πέντε φορές αναφέρθηκε η ΒΕΦΚΟ, οπότε νομίζω ότι πρέπει όντω να πω κι εγώ. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τις χώρες μέλη των χωρών μελών, είναι πιο σημαντικοί παίκτη στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου και της επιστημιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω από 8 δις έχουμε δώσει σε 60 χώρες γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ δράσει ε, σε συνεργασία με τον ΦΑΟ, με το ΙΒΑ, το με μη κυβερνητικέ οργανώσει, σε περιοχέ όπου υπάρχουν κρίσει και φυσικά υπάρχουν και ιδιωτικέ επενδύσει και θα έρθω σε αυτό αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ευχαριστεί για την έκθεση όσον αφορά την επιστημιστική ασφάλεια. Τα 790 εκατομμύρια δεν ε, μας αρέσουν είναι κάτω από ό,τι ήταν ε, πέρυσι. Πρέπει να πάμε όμως πιο γρήγορα. Η Επιτροπή έχει θέσει στόχους. Για παράδειγμα, μείωση κατά 7 εκατομμύρια των παιδιών που υποφέρουν από υποσυτισμό. Και εδώ πρέπει να κάνουμε έκκληση σε όλους και γι' αυτό στρέφομαι εδώ προς τους εταίρους μας από τη Ρώμη. Στόχους. Γιατί τότε τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να ελέγξουν κατά πόσο έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι είναι ένα κοινό μας χρέος. Αλλά ατομικά επίσης έχουμε ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε οι εταίροι μας να κάνουν περισσότερα. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα, καταπολέμηση του υποσυτισμού. Ο υποσυτισμός είναι ντροπή για τις κοινωνίες. Όχι απλώς δεν δίνουμε αρκετές βιταμίνες, ε, ε, στοιχεία κτλ. Αλλά εδώ διακυδεύεται και το μέλλον των ανθρώπων αυτών. Και δεν πρόκειται μόνο για την ποσότητα, πρόκειται και για την ποιότητα. Εκπαίδευση είναι κάτι παραπάνω από τρόφιμο, είναι θέμα πολιτιστικό. Δεύτερον, κρίση στο κέρα της Αφρικής και στο Σαχέλ. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε αντίσταση, δηλαδή πρέπει να αντέχουν οι χώρες, οι περιοχές, οι κοινότητες, οι άνθρωποι να αντιστέκονται σε φυσικές καταστροφές, σε κλιματικές αλλαγές, αλλά δυστυχώς καταστροφές γίνονται και να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους για να μπορούν να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν τις ε, καταστροφές, είτε πρόκειται για ξηρασία, είτε πρόκειται για πλημμύρες. Και επί το σχεδιασμός είναι η πρώτη μας υποχρέωση. Τρίτον, 20% του προπολογισμού μας θέλουμε να πηγαίνει σε δράσεις για τις κλιματικές αλλαγές. Το να συνδέουμε ένα ποσοστό βοήθειας σε συγκεκριμένο στόχο είναι κάτι που μπορεί να ισχύσει κι αλλού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη γεωργία που είναι θύμα αλλά και προκαλεί και κλιματικές αλλαγές κάποιοι εξέχοντες εδώ από το Κοινοβούλιο λένε ότι αν άρχισαν οι Κινέζοι να τρώνε κρέας όπως τρώμε και εμείς θα χρειαζόμασταν τρεις πλανήτες για να θρέψουμε τους Κινέζους ε, με κρέας. Θα χρειαζόμασταν γη για τα ζώα μας. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους αγρότες υπέρ της βιώσιμης γεωργίας και να γίνει καλύτερη διαχείριση της γης και του ύδατος. Γίνεται πολλή δουλειά βέβαια με την έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και να φτάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας στους αγρότες. Ήμουνα στη και στην Κένια, κοίτα πως η διοπικιλότητα και η ευπροσαρμοστικότητα βοηθούν τους αγρότες. Τέταρτον, δεν πρέπει να περιοριστούμε στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, αλλά να δούμε τη διαδικασία. Ξέρετε ότι τα απόβλητα στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι ε, μόνο μετά, είναι πριν καν φτάσουν τα προϊόντα στην αγορά. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και για να το πετύχουμε αυτό δεν φτάνει η δημόσια βοήθεια πρέπει να δώσουμε κίνητρα και για ιδιωτικές επενδύσεις. Πολύ δύσκολο όμως αυτό, γιατί οι ιδιωτικοί επενδυτές δεν πάνε εκεί που θέλουμε εμείς να πάνε, άρα πρέπει να προωθήσουμε διευκολύνσεις και πρωτοβουλίες για να βρούμε αυτές τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η γεωργία σε αναψώμενες χώρες ενισχύεται. Τέτοιες πρωτοβουλίες όμως είναι αναγκαίες αναπτύσσουμε μια νέα πρωτοβουλία που ονομάζεται AgriFi, δηλαδή είναι χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες υπέρ της Γεωργίας. Ο Επίτροπος Μιμίτσα θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία αυτή μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες στο Μιλάνο, μια που θα είσαστε κι εσείς εκεί, θα υπάρχει η διατροφική βοήθεια μεταξύ άλλων και αυτό είναι ένα θέμα που σε πολιτικό επίπεδο εδώ πρέπει να προβληθεί. Η πρωτοβουλία Γκριφάη θέλει να προωθήσει τις επενδύσεις και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο από τις μεγάλες, αλλά και τις μικρομεσαίες, γιατί αυτές είναι η σπαθολική στήλη της οικονομίας σε πολλές χώρες. Αξιότιμοι προβλευτές Όλα αυτά πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι με τις κοινωνικές δράσεις. Αναφέρθηκα πριν στην ε, παιδεία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνική προστασία. Διότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει για να αντιμετωπιστεί ο ποσιτισμός, ο οποίος έχει επιπτώσεις. Έτσι με την κοινωνική προστασία θα προωθήσουμε και την ε, παιδεία και θα μειωθεί ο ευάλωτος χαρακτήρας ε, των ανθρώπων που υποφέρουν από κοσιτισμό. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Αν δεν αλλάξουμε την κοινή κατανόηση ότι η γεωργία ε, δεν είναι ε, μία, ένα επάγγελμα που μόνο ο πλούσιο θα σας κάνει. Όχι. Δεν είναι ότι θέλουμε περισσότερη γεωργία κτλ. Αλλά πρέπει να αλλάξει το παράδειγμά μας. Η γεωργία πρέπει να μην ε, είναι αυτός σκοπός, αλλά πρέπει να βοηθάει τους αγρότες να έχουν καλύτερη ζωή και εκείνοι με τη σειρά τους να προσφέρουν σε εμάς μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό πάντα και το βλέπουμε και από την ε, μετανάστευση, εγώ σε αυτή τη μετανάστευση θα σταθώ, από την ύπεθρο της πόλης. Ακόμα υπάρχει και αυξάνεται και δείχνει ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παίζει ηγετικό ρόλο στον τομέα της διατροφικής ασφάλειας και να χρησιμοποιεί τους καλύτερους σωματοδοτικούς μηχανισμούς ώστε να πετύχουν οι στόχοι του 2030. Αλλά για να πετύχουν σημαίνει ότι όλοι, οι δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, τα κοινοβούλια, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι ειδικευμένε υπηρεσίες και οργανώσεις πρέπει να συνεργαστούν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Thank you ευχαριστούμε, λέει ο Και να αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Ο, ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής Γεωργίας, σας, παρακαλώ, μόνο ένα λεπτό παρακαλώ, λέει στον κύριο Ντοντέ. Ναι, θα να σας μιλήσω αντί του συντονιστού μας. Ήδη και επανειλημμένα το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει και σε μία τουλάχιστον έκθεση τι γίνεται με αυτά που τις τροφές που απορρίπτονται γιατί θα πρέπει κάπως να συμβάλλει η Ευρώπη όσον αφορά την ε, το πρόβλημα της διατροφής για όλο τον κόσμο. Και το G20 επίσης είπε το ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί είναι πάρα πολύ μετάβλητες οι τιμές οπότε υπάρχουν πάρα πολλές ε, χώρες σε αυτό το επίπεδο και κυρίως αυτές που είναι πιο φτωχές και ο g ανέθεσε στο, στον ΦΑΟ την αποστολή. Την αποστολή να συγκροτηθεί ένα παρατηρητήριο για να μπορεί να προβλέψει τις κρίσεις και να μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλο τον πλανήτη κάποια ελάχιστη ποσότητα ε, τροφίμων. Πώς πάνε τα πράγματα. Σικέρσκι. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε και για αυτή την ε, ευκαιρία που μας δίνεται να μιλήσουμε με τους φίλους από την ΦΑΟ. Το θέμα αυτό το, ε, το, το έθιξαν και η Επιτροπή με αυτό που είπε ο κ. Ριντόλφη, γιατί εφού υπάρχει ένα πρόβλημα κακής διατροφής, το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι ο γνώμη ότι δεν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να λύσουμε το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να θεωρήσουμε τι στρατηγικέ μα. Η κοινή γροτική πολιτική, αυτή που, που αναθεωρήσαμε κατά την περασμένη κοινοβουλευτική θητεία, ε, μας δείχνει μια σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με μια πιο πράσινη γυριά όμως, από πλευράς διαχείρισης των πόρων. Εάν η ζήτηση συνεχίσει να αυξάνει με τους σημερινούς ρυθμούς και αυξηθεί και το κατηγεφαλήν εισόδημα, τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το ότι η προσφορά δεν συνάδει προς τη ζήτηση, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια εκταρίων που χρειάζονται στην Ευρώπη. Κύριε Βαλίδη. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα αυτό πώς αντιμετωπίζουμε την σπατάλη τροφίμων. Υπάρχει όμως και η έλλειψη η ικανότητα παραγωγής τροφίμων στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες λόγω μη επαρκών υποδομών. Η Κομισιόν πάντα λέει εάν θέλουμε όλους να τους διατρέφουμε με τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά, χρειαζόμαστε τρεις πλανέτες. Μα η Ευρώπη παράλληλα έχει μια επιθετική στρατηγική εξαγωγής κρέατος, προϊόντων κρέατος. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι καλύτερα για τα θέματα αυτά και πώς ε, συνδέεται αυτό με την σπατάλη ύδατος και με την συζήτηση για την πρόσβαση στην γη, αυτό είναι ένα, ένα πραγματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα της αρπαγής γης σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό και να εξασφαλι... πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν ότι όλοι οι γεωργοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γη. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι αν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ήταν διατεθειμένη να βοηθήσει με αποφασιστικό τρόπο ώστε να λυθεί, να εκριζωθεί αυτό το πρόβλημα της ε, πείνας και της κακής διατροφής ε, θα το είχε κάνει νομίζω ότι είναι φαρισαϊκό αυτό ε, την συνείδησή μας το ότι αφιερώνουμε ε, όπως σήμερα κάποιες ε, ώρες και να μιλάμε για τη διατροφική ασφάλεια αντιθέτως οι πολιτικές ε, τις οποίες τώρα χαράσουμε παροξύνουν περισσότερο το πρόβλημα. Ήδη μίλησε ο, ο προηγούμενος συνάδελφος για το τι γίνεται με τις γέες που χάνονται, τι γίνεται με το νερό κλπ. Τι γίνεται με τις συνθήκες ελευθέρου εμπορίου. Εγώ νομίζω ότι επίσης θα έπρεπε να κάτσουμε και να αξιολογήσουμε το πώς μέσα από τις συνθήκες επιβάλλεται ότι ακριβώς εκείνες οι χώρες οι οποίες δεν μπορούν να αποφασίσουν ε, για γεωργία και για ε, διατροφή και επίσης αυτό το οποίο ε, είπανε πολλοί ότι αυτό που θέλουμε είναι το πως ναι ναι τελειώνω τελειώνω πρόεδρε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση το, αυτό που θέλει είναι να πουλήσει τρόφιμα σε αυτές τις χώρες Ένα λεπτό. Παρακαλώ να τηρείτε αυτό το χρόνο. Θυμάμαι δύο περιστασίε μου ότι είχαμε κάποιου καλόπιστου δυτικού οι οποίοι κατέστρεφαν τις δυνατότητες παραγωγής στην Αφρική. Πρώτα-πρώτα στην Ευρωδεσία. Ε, εκεί εξήγαγαν σε έξι χώρες ε, προϊόντα. Ανακατεύτηκαν ε, οι δυτικοί, φέραν τον Μουγκάμπη, ήταν σε η κυβέρνηση Σμιτ και τελικά καταστράφει παραγωγή. Επίση, κάτι άλλο που γίνεται συνέχεια είναι το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί όσον αφορά τα φυτά, τη νέα τεχνολογία. Μα αν η τεχνολογία αυτή που έχουμε εδώ για να πείσουν τα φυτά, αν το κάνουμε αυτό στην Αφρική, πολύ περισσότεροι θα είχαν πολύ περισσότερο φαΐ γιατί αφού θέλουμε να, χρησιμοποιήσουμε εκεί πέρα λιπάσματα και φάρμακα θα πρέπει εκεί πέρα βέβαια να προστατευτούν τα παιδιά, να τα μεταφέρουμε και λοιπά. Όχι δεν χρειάζεται αυτό να γίνει, δεν χρειάζονται τα λιπάσματα. Μα γιατί όλα τα κάνουμε τόσο δύσκολα για τους Να το ένα λεπτό, ένα λεπτό. Υπάρχουν πάνω από 16 εκατομμύρια άτομα τα οποία έχουν φύγει από τις χώρες τους, είναι πρόσφυγες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αντιμετωπίσει η πολιτική ανάπτυξη και τα προβλήματα των πολέμων και της προσφυγιάς. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την καταπολέμηση της πείνας είναι μια αξιοπρεπής πολιτική γεωργίας και πολιτική αλίας η οποία γίνεται με συμφωνία των χωρών όπου ασκείται και προφανώς θα πρέπει να έχουμε και μια τίμια πολιτική εμπορίου εναντί των χωρών αυτών. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να παράγουν ενέργεια. Πολλές από τις χώρες αυτές που, όπου υπάρχει πείνα δίνουν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε για την αγορά ενέργειας. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι αυτάρκεις στην ενέργεια και να μπορούν με τα δικά τους μέσα να παράγουν την ενέργεια που θέλουν. Ο Χέρμαν Σέρ έχει αγωνιστεί πάρα πολύ για την προσπάθεια αυτή α, ενεργειακής αυτάρκειας στις χώρες αυτές και είναι η πέμπτη του θανάτου του. Μπορούμε να το θυμηθούμε αυτό αύριο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί η ΦΑΟ δεν υποστηρίζει τις ε, προτάσεις του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα της ε, ΦΑΟ που μίλησε για την συμμετοχή της αγροτικής ε, των μικρών επιχειρήσεων που είναι βιώσιμες και έχουν οικολογικό χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή οι αγροτοφημικές επιχειρήσεις συμβάλλουν ιδιαίτερα σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και πρόκειται για διεθνικές εταιρείε όπως η Microsoft, η Μονσάντο και άλλες επιχειρήσεις όπως η SmithKline δεν έχουν ε, καμία μέρημνα για τις συνθήκες όπου παράγονται. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουν μεγάλες παγκόσμιες συμμαχίες. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο λέτε για τη μικρή και ευφυά γεωργία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια στροφή προς μια πραγματική ε, οικολογική γεωργία. Αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε παρά μόνο να αυξήσουμε την παραγωγικότητα των μικρών γεωργών. Καλά, εντάξει. Δεν μπορώ, δεν προφταίνω να κάνω το ερώτημα. Κύριο Άντζου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που έχουν ήδη λάβει το λόγο. Θέλω να πω ότι και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η τροποποίηση παραδείγματος στην ε, Γεωργία. Ψηφίσαμε το πρωί την αλλαγή του κανονισμού για τις βιολογικές καλλιέργειες είναι απαραίτητο να θυμίσουμε ότι η βιολογική γεωργία δεν είναι μονάχα το ότι δεν χρησιμοποιούμε παρασυντοκτόνα κτλ. αλλά ότι πρέπει να ανακτήσουμε τα εδάφη και την εφορία τους. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια σωστή εφαρμογή σε, τις γεωργικες δραστηριότητες. Πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το μοντέλο μας, πρέπει να ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκό μύθο που πιστεύει ότι εμείς έχουμε το καθήκον να ταΐσουμε τους άλλους. Αντί να σκεφτόμαστε για τους άλλους, θα ήταν χρήσιμο όταν επανέλθουμε σε μια μεταρρύθμιση της εισαγωγικής πολιτικής να σκεφτούμε από κοινού για πολιτικές όχι για τους άλλους αλλά μαζί τους με τους άλλους. Αυτή πρέπει να είναι η κυριαρχή πολιτική μας κατεύθυνση για την αγροτική πολιτική. Τσούλοφ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την ευκαιρία θέλω να κάνω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο του ΦΑΟ ή στην εκπρόσωπο. Συχνά λέμε ότι αυξάνεται ο πληθυσμός, άρα θα πρέπει να παράγουμε περισσότερα. Και έχουμε πολλές φορές ψηφίσει σύμφωνα με αυτή την αρχή. Όμως δεν συμφωνώ. Γιατί ακριβώς όπως προκύπτει από κάποιες δικές σας ε, παρεμβάσεις, ε, έτσι νομίζω ότι υπάρχει από γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να γίνει κάποια καλύτερη αναδιανομή και πιο αποτελεσματικός κύκλος παραγωγής ε, των, τροφών. Επομένως, εσείς πώς σχολιάζετε αυτή τη φράση ότι θα είμαστε περισσότεροι, άρα πρέπει να παράξουμε περισσότερα. Επόμενος, ένα λεπτό, ο Πρόεδρος. Η μεταφορά τροφίμων από τον αναπτυγμένο κόσμο προς την Αφρική, προ τον κόσμο, είναι ένα ντάμπι γιατί καταστρέφει την τοπική παραγωγή. Είναι ένα πολύ ωραίο μέτρο, κατ' επίφαση ανθρωπιστικό, που όμως είναι καταστροφικό. Έπειτα, για το θέμα της, ε, της γεών Ισραήλ, Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα κλπ. κλπ. στην Αφρική. Έχει συνέπειες να φεύγουν οι αυτόχθονες, να διώχνονται οι γεωργοί, οι περισσότεροι και αυτοί που μένουν τελικά αναγκάζονται να φύγουν εκεί Γίνεται εκμετάλλευση με τρόπο που δεν θα έπρεπε και αυτοί που νοικιάζουν τη γη προσπαθούν να αποφεληθούν όσο γίνεται περισσότερο, την εκμεταλλεύονται υπερβολικά, χάνει τις ε, θρεπτικές ουσίες και τελικά γίνεται άχρηστη. Για να μην πω για το νερό που καταστρέφεται και χάνεται πάρα πολύ πόσιμο νερό. Ο ΦΑΟ τι κάνει γι' αυτό, γιατί γι' αυτό το φαινόμενο δεν βλέπω. Ο ΦΑΟ να λέει απολύτω τίποτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μας ε, <clears throat> κάνατε να δούμε πώς η προσπάθεια, πόσο μεγάλες ήταν οι επιτυχίες για τον αγώνα κατά της ε, ε που έχουν ουσιαστικά εκμηδενιστεί από την ταχεία αύξηση του πληθυσμού. Το θέμα είναι ότι όταν μειώνεται η πείνα αυξάνεται πιο γρήγορα ο πληθυσμό σε μια χώρα ή όχι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνοδευτική κοινωνική πολιτική στις χώρες αυτές ώστε να μπορέσει να τροχοπεδηθεί αυτή η αλόγιστη αύξηση του πληθυσμού. Σκεφτόμαστε χώρες όπως το Πακιστάν, Αφγανιστάν ή Εμένη όπου μας συγκρίνουμε την κατάσταση του πληθυσμού του το 1950 και τις ε, προσδοκίες για το 2050 βλέπουμε ότι είναι τεράστια η αύξηση του πληθυσμού, επομένως δεν μπορούμε έτσι να νικήσουμε την πείνα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Χόισλινγκ. σε ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ απλό θυμάται αυτά που είπε ο Άλμπερ Άινστάιν που λέει δεν είναι απαραίτητο για να μπορέσει να επιβιώσει η ανθρωπότητα θα πρέπει να περάσει σε μια διατροφή μόνο φυτοφαγική. Η πολιτική όμως της Κομισιόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Η πολιτική αλίας μας να ενισχυθεί η πολιτική ενίσχυσε την, ε, την πείνα, η αγροτική μας πολιτική επίσης με τις επιδοτήσεις σας, η εμπορική μας πολιτική έχει αυξήσει την παγκόσμια ένδια. Είναι σαν να λέμε ωραία λόγια, αλλά τελικά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης πεινάει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις προς την Επιτροπή η κυρία Μάκαβαν και προς τους άλλους, οπότε να είστε πάρα πολύ σύντομοι όσον αφορά τις ε, απαντήσεις. Διότι σύντομα θα αποχωρήσουν στις 6.30 δερμηνείς. Ποιο θα μιλήσει πρώτο και παρακαλώ μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα μεταφράζεστε από του διερμηνεί. Ναι, ναι, θα αρχίσω και μετά πάρω την συγκεκριμένη συνάδελφη για το θέμα αυτό του, μετάβολου των τιμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όλοι ε, γνωρίζουμε και ε, την κρίση ε, του 7 με 11, αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα συγκεκριμένα δεδομένα. Ότι δηλαδή υπάρχει δηλαδή μια δύσκολη συγκυρία για την Γεωργία. Οπότε ακριβώς για τους λόγους που εξηγούν αυτή την κρίση είναι ε, το πόσα αποθέματα υπάρχουν, η πτώση του πετρελαίου, αλλά επίσης και, το, και, και, και η, οι διακυμάνσεις του δολαρίου. Βεβαίω οι χαμηλές τιμές είναι καλές για την διατροφική ασφάλεια, ε, ακριβώς επειδή υπάρχουν και απειλές για το εισόδημα που δίνουμε για να αγοράσουμε τρόφιμα. Όμως να μην ξεχνούμε ότι για να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα συνολικά. Ε, η πτώση των τιμών έχει επιπτώσεις στο εισόδημα των γεωργών. Οπότε τώρα με δύο λόγια όσον αφορά την άλλη ερώτηση για την διασπάθηση των τροφίμων νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι συνάδελφοι όταν σας ε, μίλησαν για το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματείου, το Zero Hunger Challenge, είναι ένας δεύτερος πυλώνας εκεί, ο οποίος ακριβώς αντιμετωπίζει την διασπάθηση. Ε, διότι νομίζω ότι οι χώρες τη Ευρώπη έχουν λάβει σημαντικά μέτρα πρόσφατα και ψήφισε το Κοινοβούλιο στη Γαλλία αλλά και στο Βέλγιο και αλλού ή στην Βόρεια Ευρώπη. Όμω, όμως είναι διαφορετικό το πρόβλημα στην Ευρώπη από ότι στις χώρε. χώρες γιατί το πρόβλημα σε εκείνες χώρες είναι το ότι 30 με 40% μετά τη σοδεία της παραγωγής ε, χάνεται λόγω τη κακή του, της κακής μεταφοράς τα κακών ε, συνδικών αποθήκευσης κλπ. Όλα αυτά να τα λάβετε υπόψη. Ο επόμενος κύριος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά πάρα πολύ γρήγορος, γιατί το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι μετά το, τη συνάντηση του Τζίκωση για το ευμετάλλιο των τιμών, το ΦΑΟ βρήκε άλλους και κάθισαν να τα πούνε για το Agricultural Information System. Υπάρχει τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει ακόμα και έχει πάρα πολλές πληροφορίες οπότε αρκεί τα αρχικά να τα βάλετε στο Google και θα έχετε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν και οπότε έτσι ξεκινάτε με πάρα πολλές πληροφορίες για τι γίνεται στην αγορά για, για τις τα προγνωστικά και τις τιμές κλπ. Οπότε έτσι ελπίζουμε να ανασχέσουμε αυτό το ευμετάβλητο των τιμών. Οπότε βλέπετε ότι μετά την κρίση παρακολουθήσαμε το θέμα. Οπότε τώρα με δύο λόγια να σας πω για ένα άλλο θέμα για το τι γίνεται μακρόπνα με την ζήτηση γιατί έχουμε πάρα πολλές μελέτες που μελετούν το μακρόπνον, τι προοπτικές έχει η γεωργία μακροπρόθεσμα. Οπότε είπαν ότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τα κίνητρα αύξηση της παραγωγής και ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται ορθολογιστικά και από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος. Και όχι επειδή έτσι διατάσσουν, αλλά επειδή ε, η ζωή μας οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης. Τι να, έτσι είναι η ζωή. Αλλά βέβαια μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα τα όσα έχουμε σήμερα. Αλλά αμετάκλητα θα αυξάνεται η παραγωγή όσον αφορά την συρρήκνωση της έκτασης της γης σε κάποιες περιοχές ιδίως ή στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι η ζήτηση της γης για αστικούς λόγους, για ε, ψυχολογία κλπ. μας αποστερεί τη γη από άλλες χρήσεις. Ε, γι' αυτό βλέπετε να έχουμε λιγότερη γη. Οπότε βλέπετε ότι η χρήση της γης ε, έτσι πάει σταθερά. Τα προηγούμενα 40 χρόνια θα πάει και τα επόμενα 40 σταθερά. Αλλά αυτό το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι η παραγωγή, η Οπότε ίσως μπορέσουμε να καταφέρουμε αύξηση παραγωγής χωρίς να διατράξουμε το περιβάλλον. Να, ποια είναι η πρόκληση. Οπότε ίσως μπορούμε να πετύχουμε παραπάνω αύξηση της παραγωγής και αυτό να το κάνουμε με υπεύθυνο τρόπο. Να, που είναι το δυσκολότερο. Με δύο λόγια τώρα επίσης για τον πληθυσμό. Δυστυχώς, πληθυσμός και φτώχεια είναι δύο μεταβλητές που έχουν περίπλοκη σχέση. Όταν υπάρχει φτώχεια, αυξάνεται ο πληθυσμός, δεν μειώνεται. Αυτό λέει η εμπειρία. Άρα συνήθως η φτωχή τείνουν να έχουν πολλά παιδιά. Κυρίως για τα παιδιά που θέλουν εξασφάλιση για το μέλλον, σύνταξη. Σε βοηθάνε, καλλιεργούν το φαγητό κλπ. Οπότε όταν κάπως καταπονηθεί η φτώχεια, όταν θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη παιδεία για τις γυναίκες, καλύτερες συνθήκες, τότε θεωρούμε ότι η άξιση του πληθυσμού θα επιβραδυνθεί. Και όταν βελτιωθεί η κατάσταση και για, τη διατροφή ανάλογα. Και οπότε χρειάζεται πρόοδο και ευκαιρίε για καλύτερο, μεγαλύτερο εισόδημα. Εδώ βάζω τελείω. Ευχαριστούμε πολύ. Οι πυρμηνείς θα πρέπει να φύγουν στα αγγλικά. Μπορούμε να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Μπορείτε, εντάξει, έχει καλώς.